Darf Σας παρακαλώ να καθίσετε. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση για τις ενιαίες για τους ενιαίους κανόνες και την ενιαία διαδικασία πιστοτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης και ενός ενιαίου ταμείου εξυγίανσης τραπεζών. Πρόκειται για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.